και τις δομές του ευρωπαϊκού δικαίου και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θα παραμείνει ε, νομότυπη και θα εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστέψτε με, λέει ο Πρόεδρος, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι ε, ως προερχόμενος από μια πρώην κομμουνιστική χώρα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την κατάσταση. Έχω την εντύπωση ότι είναι αντίστοιχη με αυτό που είχαμε βιώσει και εμείς στη Ρουμανία. Επιτρέψτε μου να κλείσω τη συζήτηση αυτή και να περάσω στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, που είναι η ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η συγητής είναι η κυρία Κέλλερ που έχει τον λόγο για πέντε λεπτά. Thank you very much. Today, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά η πρόσβαση στην ενέργεια είναι προαπαιτούμενο για να μορφωθούν για να καταπολεμηθεί η φτώχεια στην οποία ζουν. Και άρα θα πρέπει να υπάρξει καθολική πρόσβαση στην ενέργεια, ίση πρόσβαση που θα γεφυρώνει το κενό μεταξύ πόλεων και υπαίθρου και σε λογικές τιμέ. Επίσης, για να αναπτυχθεί μια χώρα θα πρέπει ε, να έχει σταθερή πηγή ενέργειας και βεβαίως η πιο αξιόπιστη είναι αποκεντρωμένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Αλλά πρέπει και η παραγωγή να λαμβάνει υπόψη άλλα ζητήματα όπω την κλιματική αλλαγή, την αποδάσωση, την υποβάθμιση του περιβάλλοντο, την ανθρώπινη υγεία και την φτώχεια που προκαλεί. Τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ορυκτά καύσιμα. Τα ορυκτά καύσιμα έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για την υγεία, το περιβάλλον και το κλίμα. Ταυτόχρονα, η κλιματική κρίση προκαλεί περισσότερη ζημιά σε όσους ζουν σε ακραία φτώχεια τα ορυκτά καύσιμα δημιουργούν ρήπανση που ε, θέτει σε κίνδυνο και την ανθρώπινη υγεία και την υγεία του περιβάλλοντος είναι ακριβά και η τιμή τους αυξάνεται όσο εξαντλούνται. Τα ορυκτά καύσιμα δημιουργούν κεντρικές δομές διανομής της ενέργειας. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να βοηθήσουμε τις αναψώμενες χώρες να μην περάσουν από το δικό μας το στάδιο των ορυκτών καυσίμων. Μόνο οι ανανεώσιμες μπορούν να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν θα εξελιχθούν ποτέ και πολλές αναψώμενες χώρες έχουν σε αυθονία ήλιο και αέρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τοπικά σε μικρή και φτηνή κλίμακα που ε, θα βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο να δοθεί ισχύ σε αυτούς τους ανθρώπους. Η αποκεντρωμένη ενέργεια είναι δημοκρατική στα χέρια των ανθρώπων. Όμω η Παγκόσμια Τράπεζα εξακολουθεί να προωθεί στην ενεργειακή στρατηγική τη τα ορυκτά καύσιμα. Οι πρόσφατε αυξήσει για τα δάνεια για τις ΑΠΕ παραμένουν μικρές και δεν καλύπτουν τις προφανείς προτιμήσεις. Επίσης, οι επενδύσει αυτές λαμβάνουν χώρα και μέσω ενδιαμέσων, που δεν επιτηρεί επαρκώς η Παγκόσμια Τράπεζα. Η τράπεζα εξακολουθεί να κάνει σημαντικές επενδύσεις ε, σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από άνθρακα και άρα δεσμεύει αυτές τις χώρες για δεκαετίες. Δεν είναι έτσι η ενεργειακή επανάσταση. Η ενεργειακή πολιτική της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι αδιαφανής και το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω του ορισμού ξεκάθαρων απαιτήσεων που θα πρέπει να εκπληρώσουν η οικονομική ενδιάμεση για να έχουν πολυμερή χρηματοδότηση. 40% των δανείων της Παγκόσμιας Τράπεζας στον ιδιωτικό τομέα πηγαίνουν μέσω αυτών των ενδιαμέσων και μεγάλο μέρος αυτών των δανείων πηγαίνει στον τομέα της ενέργειας ιδιαίτερα Όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες ε, διαθέσιμες για τα προϊόντα αυτά τα επενδυτικά και δεν μπορούμε τελικά να δούμε το τι συμβαίνει στη χρηματοδότηση των ενδιαμέσων. Και αν δούμε το τι ενέργεια θεωρούν χαμηλού άνθρακα, βλέπουμε μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τόσο μεγάλα που καταστρέφουν μεγάλο μέρος της ε, φύσης και διώχνουν ανθρώπους από τα σπίτια τους. Δεν είναι αηφόρο αυτό και δεν είναι προς ε, το συμφέρον ε, των ανθρώπων και της κοινωνίας. Επίσης, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακας δεν, άνθρακα δεν κάνει τον άνθρακα χαμηλού χαμηλή ένταση. Το διοξείδιο του άνθρακα ακολουθεί να υπάρχει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει ε, κάτω από τη γη. Κανείς δεν μπορεί να πει πως θα παραμείνει εκεί πέρα ήρεμα για τις επόμενες χιλιετίες. Αυτό είναι μαντία και όχι έρευνα. Και οπωσδήποτε όχι πολιτική. Το ίδιο ισχύει για την πυρηνική ενέργεια. Η εξόριξη ουρανίου παράγει τεράστιε ποσότητες διοξείδιου του άνθρακα και κανεί δεν ξέρει τι να κάνει με τα απόβλητα. Αυτό δεν είναι αϊφόρο και χαμηλού άνθρακα. Γι' αυτό οι πράσινοι καταψηφίζουν το ψήφισμα ε, εκτός αν αντικατασταθεί η διατύπωση για το χαμηλό άνθρακα. Όμως υπάρχουν και ορισμένα καλά στο ψήφισμα, όπω παραδείγματο χάρη η εστίαση σε ανανεώσιμες εκτός δικτύου για μικρής ε, έκτασης παραγωγή και όχι τα μεγάλης κλίμακας εργοστάσια για εξαγωγή βιοκαυσίμων. Επίσης, το κόστος της μεταφοράς τεχνολογίας και ειδικά η μεταφορά τεχνολογίας δεν θα έχει πάρα πολύ νόημα εάν τηρηθούν τα πνευματικά δικαιώματα. Ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι να συμπεριφερθούμε στα δικαιώματα αυτά με τρόπο ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε λογικές τιμές για την ε, αυτό υποσχεθήκαμε στις διαπραγματεύσεις ε, για το κλίμα και ε, πρέπει να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεσή μας. Δέχεστε ερώτηση από τον κύριο Μάρτιν, κυρία Κέλλερ. Παρακαλώ κύριε Μάρτιν. 30 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μπορώ να σας συγχαρώ για αυτά τα οποία είπατε, για την ανάλυση σας. Το ερώτημα είναι, τα προβλήματα αυτά τα ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχει επειδή το έχετε δει το ζήτημα αυτό σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, υπάρχει κάτι το οποίο σας κάνει αισιόδοξη για την ε, πρόοδο της Παγκόσμιας Τράπεζας, εάν πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Όντω ε, συζητάμε τα θέματα αυτά πλέον των 20 ετών και ελπίζω πραγματικά ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα μάθει κάτι από τις συζητήσει αυτές, γιατί όλοι πλέον συμφωνούν ότι το μέλλον βρίσκεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είδαμε μια μικρή αλλαγή στρατηγική αυτή που είναι κάπως στρέφεται προς τι ανανεώσιμες, αλλά αυτό το μικρό βήμα πόρο απέχει του επιθυμητού, υπάρχει η απόλυτη κυριαρχία των ορεικτών καυσίμων και η υπερβολική εστίαση στους ε, υδροελεκτρικού σταθμούς που δεν είναι ούτε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ούτε βιώσιμη οποιονδήποτε. Ελπίζω λοιπόν το κοινοβούλιο αυτό να εκφράσει στεναρά και με σαφήνεια την θέση του ότι θέλουμε πραγματικά πολιτική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ευελπιστώ να, να βγάλουμε την έκφραση χαμηλής εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα και να πάμε σε σωστή χρήση και εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κέλλερ. Και τώρα το λόγο έχετε εσείς, κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είχα κάνει κι εγώ μια πολύ ισχυρή δήλωση και τονίζω καταρχά ότι η ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμια Τράπεζα είναι ευπρόσδεκτη γιατί η Παγκοσμία Τράπεζα διαδραματίζει πολύ ιδιαίτερο ρόλο στον κόσμο και δει σε θέματα αναπτυξιακά. Δεν ε, είναι, δεν είναι ο χειρισμός να πούμε ότι είναι πραγματικά ηγέτες σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές στρατηγικές. Καταρχάς λοιπόν τονίζω ότι όντω πρέπει με απόλυτη σοβαρότητα να δούμε το θέμα του ρόλου τη παγκόσμια τράπεζα και τη ενεργειακή στρατηγικής τη. Ταυτόχρονα όμω, υπάρχουν και κάποια ζωτική σημασία θέματα όταν ε, αποτιμούμε την δική μα ανταπόκριση στρατηγική αυτή. Στρατηγική αυτή. Εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιο αριθμό νοικοκυριών που δεν έχουν καμία απολύτως πρόσβαση σε οποιαδήποτε τύπου ενέργεια. Και είναι αλήθεια ότι 20 χρόνια συζητάμε το ίδιο θέμα. Όμω, πολύ σημαντικές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα ή γενικά στην παροχή υπηρεσιών ενέργειας δεν έχουν τελικά αποδώσει για εκατοντάδες εκατομμυρίων ατόμων, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς νοτίως της Σαχάρας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει καταρχάς να κατανοήσουμε την κλίμακα της πρόκλησης. Το δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι το θέμα της ε, ανάπτυξης. Κάθε μία από τις χώρες αυτές που είναι στην πορεία προς την ανάπτυξη έχουν τεράστια ζήτηση και το μέγεθος της ζήτησης θα πρέπει να, να καλυφθεί με την αντίστοιχη παροχή. Άρα αυτό δίνει, αν θέλετε, το πλήρω της όλης κλίμακας. Και τρίτο και συμφωνώ απόλυτα είναι το θέμα της αηφορίας και της προσμονής. Οτιδήποτε και να κάνει ο ενεργειακό τομέα, θα πρέπει να δούμε και ποιε θα είναι οι συνέπειε και οι επιπτώσει στην κλιματική αλλαγή. Και ξέρουμε ότι ο υφιστάμενος ενεργειακό τομέα προκαλεί το φαινόμενο θερμοκηπίου. Και επίση θα πρέπει να εξετούμε και ποιε είναι οι τιμέ των ρηκτών καυσίμων. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η πρόκληση των τιμών την ορυκτών καυσίμων είναι μπροστά μας. Και ελπίζω ότι θα το δούμε το θέμα του στο του δυνατό, αλλά είναι αναπόσπαστο κομμάτι, αν θέλετε, της σχεδιασμού, της προσμονής επόμενης στρατηγικής. Θα ήθελα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μελετήσει πραγματικά το πράσινη χάρτα για την όλο προσανατολισμό που έχουμε δει σε ό,τι αφορά το ενεργειακό τομέα, όπου έχουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες ως έναν κεντρικό πυλώνα των νέων κοινοτικών πολιτικών. Γιατί εάν δεν κάνουμε αυτό το πρωτοπόρο πείραμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιμένουμε, αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, ότι μπορούμε να πείσουμε την Παγκόσμια Τράπεζα, οποιοδήποτε άλλο φορέα, ότι θα πρέπει να εστιάσουμε τις επενδύσεις μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να έχουμε το θάρρος για κάτι τέτοιο. Απαιτούνται πάρα πολλά, πάρα πολλοί χρηματοοικονομικοί πόρη στις μέρες μας για να μεταστραφούμε σε αυτό το τομέα. Απαιτούνται αρχικά πολύ ψηλέ επενδύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά βλέποντας πώς κοιμώνονται κυμαίνονται και πώς θα κινηθούν οι τιμές ενέργειας, σίγουρα οι ανανεώσιμες είναι οι προτιμητές ό,τι αφορά το μέλλον. Και η γνώση μας η σημερινή μας δίνεται έγκυα ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε πολύ μεγάλη αλλαγή σε αναπτυσσόμενες χώρες και πιστεύω ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό. Ξέρω ότι η υδροηλεκτρική, η υδροηλεκτρικός τομέας είναι ένας προκλητικός τομέας, αν θέλετε, από κάθε άψη. Αλλά σε ό,τι αφορά τις αναλύσεις βιωσιμότητας, νομίζω ότι είναι πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα γιατί οι περισσότερες χώρες έχουν τεράστια ισχύ μέσα των υδάτων. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση και συζητήσουμε τα θέματα της πολιτικής, της πράσινης χάρτας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν υπέρ της, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εάν επιμέναμε και αν ενισχύσετε αυτή την, την πράσινη χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπορούσαμε να πείσουμε και τρίτους και δει την Παγκόσμια Τράπεζα, ώστε να εστιάσουν περισσότερο στους ε, σταθμούς ε, ε μικτής παραγωγής. Υπάρχουν έξι βασικά κριτήρια για τις μελλοντικέ επενδύσεις. Η Παγκόσμια Τράπεζα υπό τον Bob Σόλοκ είναι εξαιρετικά δραστήρια και ενεργή στις όλες τις συζητήσεις. Το ότι συμμετέχει λοιπόν εργά η Παγκόσμια Τράπεζα είναι κάτι υπέρ δεν πρέπει να το φοβόμαστε, είναι σύμμαχος, αλλά πρέπει όμως να υπάρχει η ευρωπαϊκή ηγεσία στο τομέα αυτό. Δηλαδή στον ενεργειακό τομέα για, τις αναπτυσσό... για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ένα άλλο θέμα το οποίο τέθη, και είναι στο ερώτημα, αφορά τον ΠΟΕ. Η Συμφωνία Κοτονού είναι είναι, ε, είναι βασικό μέσο μαζί με την, ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την χρηματοδότηση υποδομών για προγράμματα ήπια και φιλικά προς το περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα, δεν υφίστανται ειδικά σχέδια στο πεδίο των αρρυκτών καυσίμων. Η γενική πολιτική είναι σαφέστατη. Χρηματοδοτούμε ενεργειακά προγράμματα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, που βασίζονται είτε στην πράσινη ενέργεια, είτε την αιωλική, είτε την ηλιακή. Στα πλαίσια της ενδιάμεσης έκθεσης που καλύπτει τις χώρες Ασίας, ε, Λατινικής Αμερικής και Νοτιού Αφρικής, ε, προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργοποιηθούν επιπρόσθετα δύο δις για το 2011-2013 για να υποστηριχθεί οι σχετικές χρηματοδοτούμενες διαδικασίες μέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων στο πεδίο της, ε, ε απάλυνσης του φαινόμενου του θερμοκηπίου και της προαγωγής φιλικών μορφών ενέργειας. Έτσι λοιπόν περιλαμβάνονται οι απαραίτητες διατάξεις ώστε μόνο έργα τα οποία είναι οικονομικά, κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά η φόρα θα υποστηρίζονται κάτω από την εντολή αυτή που έχει δοθεί στην ε, ΕΤΕ. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα βήματα για να, δίνουμε, να λάβουμε ηγετικό ρόλο στον κόσμο στο πεδίο αυτό και για να ε, κατευθύνουμε και τη σχετική ενεργειακή πολιτική της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θέλουμε λοιπόν τώρα να δώσουμε το λόγο στους ε, ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Εκ μέρους του ΕΛΚ, λοιπόν. Ο κύριος Σβένσον. Για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Εκτός μικροχώνου. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό που βρίσκεστε ε, εδώ, παρόλο που ο χρόνος που έχουμε δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιος. για τα ορυκτά κάψιμα, μιλήσατε για τις επενδύσεις και για την Παγκόσμια Τράπεζα που έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και μιλήσαμε και για την τακτική της ε, παροχής ε, κινήτρων Πρέπει όμως να δούμε πως θα εφαρμοστούν στην πράξη αυτά τα διάφορα έργα και μην ξεχνάτε, γιατί εσείς είπατε ότι υπάρχουν δυνατότητες να δράσει σε πρακτικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο, στην Αφρική, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική. Νομίζω όμως, κύριε Πρόεδρε, γιατί τον, τον έχω ακούσει πολύ συχνά να μιλά για το σημείο αυτό τον Επίτροπο, πως Έχουμε πολλούς ε, πρόωρους θανάτους επειδή πολλά νοικοκυριά δεν έχουν τους πόρους για να επιβιώσουν. Αυτό συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη αυτά να ε, επενδύουν σε ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες ή σε ε, συστήματα συλλογής ηλεκτρικής ενέργειας, σε θερμοσυσσωρευτές. Καλό είναι λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιου είδους project. Να μην χρησιμοποιούμε λοιπόν ε, τα ξύλα του που προέρχονται από την υλοτομία, όταν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά ας το περιγράψουμε με όρους πρακτικούς, να προτείνουμε κάποιες εναλλακτικέ λύσεις και να πούμε πως εκτός από την ελληνική, την ολική ενέργεια και την ηλική ενέργεια υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Επαναλαμβάνω λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε στην πράξη ποιες δυνατότητες υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή Ήδη έχουμε καθυστερήσει και εμείς θα έπρεπε να είμαστε η αιχμή του δώρατο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντικαταστήσουμε αυτά τα ορυκτά καύσιμα με κάτι διαφορετικό και εμείς και ο αναπτυσσόμενος κόσμος. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των σοσιαλιστών. Ο κύριος Πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Πίμπαλς, καταρχήν να συγχαρώ τη Σκά Κέλλερ για την εξαιρετική δουλειά της στην έκθεση αυτή πραγματικά όσοι δουλέψανε σε αυτή την έκθεση είδαν ε, το πόσο μη βιώσιμη είναι από πολλές πλευρές η στρατηγική της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας. Πόσο, όπως είπε και η Σκά το ότι μεγάλα έργα, έργα μεγάλης κλίμακας, μη βιώσιμα, όπως τα υδροελεκτρικά και πολλά άλλα. Είναι όντως γεγονός ότι αυξήθηκε κατά 300% η χρηματοδότηση για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. την ίδια στιγμή όμω Επίτροπη αυξήθηκε και 430% η χρηματοδότηση των έργων ε, ορυκτών καυσίμων fossil fuels. η παγκόσμια τράπεζα και αυτό είναι θα έλεγα σκανδαλώδε, δεν υπολογίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των έργων που χρηματοδοτεί η ίδια. την ίδια στιγμή ακόμα και σήμερα συζητά την της χρηματοδότηση. Ε, project που αφορούν ε, palm oil plantations φυτείες ε, φινικέλαιου. δεν σέβεται τις αρχές της ελεύθερης και πρώτερης και μετά από επαρκή πληροφόρηση συμφωνίας των Ιθαγενών για τα έργα που χρηματοδοτεί. είναι η αρχή του free prior informed consent. επίσης δεν ενσωματώνει και θα πρέπει να ενσωματώσει το full cycle ανάλυση το κόστος για τη ζωή, για το κύκλο ζωής των έργων τα οποία χρηματοδοτεί. Ελπίζω πραγματικά αυτή η έκθεση, όπως θα προκύψει μετά τελική ψηφοφορία, να στείλει ένα δυνατό μήνυμα ε, για τις απαραίτητες περιβαλλοντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ε, ολοκληρώσει η Παγκόσμια Τράπεζα στο εσωτερικό της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γκέρεντς, εκ μέρους των φιλελευθέρων. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η Παγκόσμια Τράπεζα, λόγω της εντολής που έχει, έχει ως στόχο την εξάλληψη της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα project να έχουν τον ίδιο στόχο. Να παρεύουν στον κοινωνικό τομέα και να προκρίνουν project τα οποία θα προσφέρουν πόσιμο νερό, σχολεία, όλα αυτά που θα μας βοηθήσουν ως προτεραιότητα να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, επαναλαμβάνω σύμφωνα με την εντολή που έχουμε δώσει αυτή την τράπεζα. Στην προφορική ερώτηση την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή, που εκφράζονται πολύ έντονες ανησυχίες για την χρηματοδότηση project ε, πετρελαϊκών ή ενεργειακών ε, που βασίζονται σε κατανάλωση άνθρακα, έχω να πω το εξή. Καταρχήν, στην ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει να έχουμε κριτήρια αξιολόγησης αυτών των έργων. Δηλαδή, να ξέρουμε πώς μπορούμε αυτά τα οποία αξιολογούμε και πώς τα κριτήρια αυτά της αξιολόγησης ε, θα λαμβάνονται υπόψη αυτήν την εκκίνηση κάποιο έργο. Θα πρέπει η με Τράπεζα και οι εταίροι της να λάβουν υπόψη και την οικονομική διακυβέρνηση των χωρών που δανείζονται. Προώθηση επίσης των ΑΠΕ ε, σε ένα κόστος λογικό που θα προκρίνει τη χρήση τέτοιου είδους ενέργειας. Και ένα στοιχείο στο οποίο ήδη έχει απαντήσει ο Επίτροπος, αλλά είναι κάτι το οποίο εμάς μας ανησυχεί ιδιαίτερα, είναι η ΕΤΕ από πλευρά της θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ε, παραπάνω παρατηρήσεις που έκανα. Επιθυμώ λοιπόν, εύχομαι λοιπόν η Παγκόσμια Τράπεζα να ενστερνιστεί αυτές τις ε, ανησυχίες και τις επιθυμίες τις οποίες εκφράσαμε εμείς εδώ και μια και τα 27 κράτη-μέλη είναι επίσης ε, εκτός από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας πρέπει με κάποιο τρόπο να επηρεάσουμε και εμείς την πολιτική αυτής της υπηρεσίας. Θα μπορούσε λοιπόν και εκεί ε, να γίνει μια συζήτηση για τα κριτήρια τα οποία τυπώσαμε και ευχαριστώ και πάλι την κυρία Κέλλερ για την εξωτερική δουλειά που έκανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι η Μαρίζα Ματίας για 2,5 λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω πως ε, εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά των ε, συναδέλφων ε, και συμφωνώ πλήρως με αυτά τα οποία ακούστηκαν. Το θέμα για το θέμα αυτό θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση που πιστεύω πως αξίζει να ακουστεί. Έχουμε μια σειρά εγγράφων ε, τα οποία δεν έχουμε ακόμα συζητήσει. Έχουμε ψήφισμα και πολλά άλλα τα οποία αφορούν το τι χρηματοδοτεί η Παγκόσμια Τράπεζα, το τι πρέπει να προωθηθεί στην Ήπεθρο και το πόσο λίγοι ε, επιτυχία υπάρχει. Η πιθανή αλλαγή ενεργειακής στρατηγικής της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2011 προβλέπεται, αλλά ε, δεν ξέρουμε εάν θα συμβεί όντω. Οπότε το θέμα μας εδώ πέρα είναι πράγματι η καταπολέμηση της φτώχειας και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά και η κλιματική αλλαγή πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ε, τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν ε, όμως να ορίζουν την ενεργειακή στρατηγική της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. έχουμε ώρες ώρες την εντύπωση πως ε, μέχρι ε, πως για μια σειρά ετών θα υπάρχει χρηματοδότηση για τα ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το πώς ε, θα χρηματοδοτήσει και πιο μικρής κλίμακας έργα η Παγκόσμια Τράπεζα και όπως είπα να λάβει υπόψη τη ναι, κλιματική αλλαγή. Οπότε το όσον αφορά το πρώτο ερώτημα γιατί δεν έχουμε ένα σωστό συμπέρασμα γιατί επιτρέπουμε αυτός ο οποίος πληρώνει να αποφασίζει κιόλα. γιατί αποφασίζουμε, γιατί αποφασίζει εδώ πέρα η ε, Παγκόσμια Τράπεζα την ενεργειακή ε, στρατηγική του κόσμου. Αν λάβουμε εμείς μία απόφαση, ε, θεωρώ πως πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Και γιατί ε, θέλουμε μια ενεργειακή στρατηγική να την επιβάλλουμε στις υπόλοιπες χώρες όταν μπορεί να μην τους ταιριάζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χάνς Πέτερ Μάρτιν έχει το λόγο τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη δεκαετία του 70, αρχή, αρχές του 80, η οικολογική τύφλωση της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας ήταν μεγάλο θέμα. Και τότε ακούγαμε τους ίδιους λόγους όπως και σήμερα. Και υποσχέσεις από την Παγκόσμια Τράπεζα. Και λέγαμε πώς θα αναμορφωθεί η Παγκόσμια Τράπεζα. Πέρασαν δεκαετίες. Και έχουν υπάρξει πάρα πολλά έργα σε πάρα πολλέ χώρες από τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες. Πού είναι λοιπόν όλα αυτά τα έργα, πού είναι τα, οι εγκαταστασει εγκαταστάσεις, πού είναι ε, η, τα δάση, τα υφόρα στον Αμαζόνιο ή αλλού, πού είναι τα ηλιακά πάνελ ε, και οι ανεμογεννήτριες στην Κένια. Τίποτα. έγινε το σύστημα το οποίο έχουν αντιγράψει πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτοδιαχείριση έπεσαν στα χέρια των μεγάλων συμφερόντων και δεν έγινε τίποτα. Και είναι απεγνωσμένοι οι άνθρωποι από τον τρίτο κόσμο και απορούμε που λένε δεν θέλω να ζω στην Καραϊβική, θα πάω στην Αμερική. Ε, απορούμε μετά που έρχονται όλοι από το Μαγκρέμπ σε εμά. Υπάρχει μεγάλη υποκρισία εδώ πέρα και βλέπετε η ριζοσπαστικοποίηση αυτών των εκατομμύριων ανθρώπων σημαίνει πως φτάνει. Και όποιος δει αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να πει δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να μιλήσουμε με πιο δυνατή φωνή και να ζητήσουμε από την Παγκόσμια Τράπεζα να κάνει κάτι. Τι κάνουν όλες οι επιτροπές εδώ πέρα, Επιτροπή Ανάπτυξης, ΑΚΕ, αν το αποτέλεσμα είναι ένα κομματάκι χαρτί, το οποίο, με συγχωρείτε δηλαδή, είναι τα ίδια συμπεράσματα που βγάζαμε στη δεκαετία του 70. Είναι πραγματικά, προκαλεί πραγματικά ντροπή. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε λοιπόν με τις πολιτικές ομάδες και τώρα θα περάσουμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Πρώτος ο κύριος Κατσμάρκ για δύο λεπτά. Στα κύριε Πρόεδρε. Σήμερα κανείς δεν αγνοεί τη σημασία της ενέργειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατ' επανάληψη υπήρξα μάρτυρας της ε, ε, έκπληξης ατόμων όταν μάθανα την τιμή ενεργειακής μονάδας στην Αφρική. Νομίζω ότι η Παγκόσμια Τράπεζα ε, έχει τεράστιο ρόλο στον ενεργειακή ανάπτυξη των απτυσσόμενων χωρών. Η ο, πολιτική μου ομάδα ζήτησε ξεχωριστή ψηφοφορία επί του θέματος. Πιστεύουμε ότι σε κάποια σημεία το ψήφισμα είναι εξαιρετικά επικριτικό απέναντι στην Παγκόσμια Τράπεζα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να απευθύνουμε παρατηρήσει στην Παγκόσμια Τράπεζα για το ποιε είναι καθαρέ πηγέ ενέργεια ή όχι, ή ποιε είναι επιθυμητέ ή όχι. Δεν νομίζω ότι είναι θεμητό. Η πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιείται κατά κόρον στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες οι οποίες εξαρτώνται από το κάρβονο και το φυσικό ε, αέριο, ε, αν θέλετε, επιπλήττονται γιατί πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές του διοξείδου του άνθρακα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να υποδείξουμε σε, εξωτερικά, σε εξωτερικές χώρες τι είδους ενέργεια επιτρέπεται να αναπτύξουν. Από την άλλη, συμφωνούμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα τα τοπικά σχέδια μικρή κλίμακα, σχέδια δηλαδή με χαμηλέ εκπομπέ. Να προάγουμε τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών για ακριβώ να μην υπάρξει εξάρτηση. Θέλουμε η Παγκόσμια Τράπεζα να επενδύσει σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και στη μεγαλύτερη, πιο αποτελεσματική χρήση τη ενέργεια. Πρέπει να έχουμε κατά νου το κύριο στόχο Δηλαδή σε ποιο βαθμό η πρόσβαση στην ενέργεια μπορεί να επιτρέψει στους λαούς να βγουν από τη φτώχεια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, να επιτύχουμε σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Να μειώσουμε τις εκπομπές, να λάβουμε υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, τα νέα, περιβαλλοντικά, στα νέα ε, σχέδια, τα ενεργητικά και να αυξήσουμε την, ε, το διαθέσιμη ενέργεια και την ε, παραγωγή ενέργειας να αναπτυσσόμενες χώρες. Ξέρω ότι ο, ο Επίτροπος δεν δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό. Τίθεται ζήτημα της πράσινη ε, χάρτας και το Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει την όλη στρατηγική. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα δίνουμε το λόγο στην κυρία Σίλβια Τσικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε αυτή τη στιγμή 1,4 δις στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στον ηλεκτροτουρισμό, από τον οποίο το 85% σε αγροτικές περιοχές. Επομένως, ε, είναι πολύ σημαντικό σημείο πρόοδου για να υπάρχει πρόσβαση, για να επιτευχθούν οι στόχοι της ε, χιλιετίας, γιατί έθεσαν, έθεταν ακριβώς τον στόχο αυτό για να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Αλλά για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να πούμε ότι περίπου 400 εκατομμύρια ανθρώπων θα έχουν πρόσβαση και περίπου ένα δις θα έχουν πρόσβαση σε ε, παρασκευή τροφής κατά τηρώντας κάποιους κανόνες υγιεινής. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχουν 0,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ να διατεθεί για κάτι τέτοιο. Η πρόσβαση ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι ο πιο σημαντικός στόχος. Ανάμεσα στα εμπόδια που οποία έχουν γνωριστεί για τον εξηλεκτρισμό των χωρών αυτών είναι μεταξύ άλλων το πολύ υψηλό κόστος για την ε, παροχή ηλεκτρισμού στις αγροτικές περιοχές και τα προάστια, η πολύ χαμηλό δυναμικό ανάπτυξης και προγραμμάτων εξηλεκτρισμού στις χώρες αυτές, καθώς και η περιορισμένη δυνατότητα ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αγροτικές περιοχές έχουν διαφορετικά προβλήματα. Σε αυτές τις ζώνες όχι μόνο πρέπει να εξασφαλιστεί απαραίτητη ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα η διαδικασία παραγωγής ε, ηλεκτρισμού δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ε, θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Ε, η Παγκόσμια Τράπεζα σε πρόσφατη έκθεσή τη, έδειχνε ότι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια αν χορηγηθούν σε προσιτή τιμή είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα, πολύ πιο μακροπρόθεσμες οικονομικά. Και αυτή η παραγωγή ενέργειας μπορεί να έχει πολύ σημαντικό ρόλο και στην εξασφάλιση ενεργειακής ανεξαρτησίας των χωρών αυτών. Αυτή η παραγωγή μπορεί να μειώσει τις εισαγωγικέ και να ε, αντιπαλέψει την πολύ μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών σε πετρέλαιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να υποστηρίξει ένα σχέδιο το οποίο στοχεύει στην εξοικονόμηση και καλύτερη χρήση του ενεργειακού αποθεματικού, θα πρέπει να στοχεύει στην εκμετάλλευση τοπικού ενεργειακού δυναμικού και να διασφαλίσει και τη διασύνδεση μεταξύ διαφόρων χωρών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, επόμενος ομιλητής, κ. Μπαλσίτης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για μια ερώτηση η οποία είναι πολύ επίκαιρη και βέβαια πολύ ενδιαφέρουσα. Η ενεργειακή ένδυα είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό και δεν επιτρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του αναπτυσσόμενου κόσμου, οι συνθήκες διαβίωσης. Μειώνει τις δυνατότητες που έχουν ε, την οικονομική ανάπτυξη και αυτά είναι ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία δεν επιτρέπουν οι χώρες αυτές να ανθίσουν οικονομικά. Ε, παραμένουν με τον τρόπο αυτό στη φτώχεια. Τα στατιστικά δεδομένα είναι πολύ ανισχυτικά. 1,5 δις ε, ανθρώπων δεν έχουν πρόσβαση ηλεκτρική ενέργεια. 1,7 δις ανθρώπων ε, χρησιμοποιούν ακόμα ε, καύσιμα βιολογικά και δύο εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της χρήσης αυτών των καυσίμων. Άρα λοιπόν τα έργα της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν έχουν δώσει ακόμα απτά αποτελέσματα και τα ορυκτά καύσιμα είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις για τις μονάδες ε, θερμοελεκτρικής παραγωγής ενέργειας. Ε, Αυτή είναι η μεγάλη ρηπαίνοντες και η συμφωνία στην G20 της μείωσης των ε, έργων που ε, βασίζονται στη χρήση ορεικτών ε, καυσίμων και το γεγονός πως θα καταργηθεί η χρηματοδότηση αυτών από το 2015 και μετά είναι ένα βήμα το οποίο κρίνεται πολύ θετικά. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τον έλεγχο και την εποπτεία στο σημείο αυτό έτσι ώστε τα έργα αυτά να συνεισφέρουν στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτών των ανθρώπων όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητά μέλη. Ε, φτάνουμε προς το τέλος της ε, σημερινής Ολομέλειας. Περνάμε λοιπόν τώρα ε, στη διαδικασία Catch the Eye. Κύριε Ρούμπικ, σε ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Επίτροπο Πίμπαλξ ως πρώην Επίτροπος Ενέργειας γνωρίζει τα της ε, στρατηγικής μας και ελπίζω η αναπτυξιακή συνεργασία να προχωρήσει περισσότερο είτε μιλάμε για τεχνική αρρωγή γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να πληρώνει μόνο στην Παγκόσμια Τράπεζα, δεν μπορεί να είναι μόνο payer αλλά να γίνει και player ο ενισχυμένος ρόλος της Ευρώπης ε, στην Παγκόσμια Τράπεζα θα αποτελέσει βασική πρόκληση για να δούμε πώς θα μπορέσουμε με την αναπτυξιακή βοήθεια να ενισχύσουμε οικογενειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην παραγωγή ενέργειας, γιατί πολλές μικρές επιχειρήσεις ε, τελικά αν τις προσθέσουμε μαζί είναι οικονομίες κλίμακας και μπορούν να προσφέρουν απόδοση στην επένδυσή μας. Επίσης σημαντικό θέμα είναι η αποθήκευση της ενέργειας και αυτό θα παίξει με σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σον Κέλλη έχει τώρα τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι είμαστε εδώ πέρα τέτοια ώρα, Μάλλον έχουμε κάποια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που μας παρακινεί. Δεν ξέρω. Ίσως και θεία χάρη την να βρισκόμαστε εδώ. surprisingly because... η συζήτηση ήταν ε, πολύ ποικιλή και λογικό δεδομένο του θέματος. Ε, σωστά, ο κύριος Επίτροπος νομίζω βρήκε την ισορροπία για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Κάποια πράγματα πρέπει να τονιστούν. Πρώτα απ' όλα, οι χώρες εάν είναι στον αναπτυσσόμενο είτε στον ε, ανεπτυγμένο χώρο, εάν έχουν πόρους, οι όποιοι και αν αυτοί θα τους χρησιμοποιήσουν. Το θέμα είναι εάν τους χρηματοδοτούμε ή όχι. Προφανώς στην Ευρώπη, από πλευράς Κανκούν και τα λοιπά, θέλουμε να προωθήσουμε εμείς ε, τις ΑΠΕ και αυτό είναι σωστό. Και ο κύριος Μάρτιν έχει δίκιο κατά μία έννοια. Ε, πρέπει να μιλήσουμε με δυνατό τρυφωνή και να σπρώξουμε την Παγκόσμια Τράπεζα για να προωθήσει περισσότερα έργα ανανεώσιμων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος ο Επίτροπος Πίμπαλξ έχει το λόγο. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό η συζήτησή μας, ακόμα και τόσο αργά, διότι η ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι μια ευκαιρία. Είναι πραγματική ευκαιρία να ανταποκριθούμε στις ενεργειακές προκλήσεις. Αν δούμε τι λέει και η Διεθνής ε, ε, Υπηρεσία Ενέργειας σε ό,τι αφορά το δυναμικό, το ενεργειακό δυναμικό και της ανώσπλης ενέργεια είναι τεράστιο το δικαιωμένο. Η Παγκόσμια Τράπεζα με τη σωστή καθοδήγηση μπορεί να επιφέρει τις απαραίτητες ε, αλλαγές. Μιλούσαμε για τον στόχο των ανεώσιμων πηγών ενέργεια που είχε θεσπιστεί, που φαινόταν έστω και ταπεινό πω ήταν την εποχή εκείνη και μετριοπαθή ο στόχο. Εν τούτη φάνηκε ότι ε, ήταν ανέφικτο τότε. Τώρα όμω φαίνεται με σωστή πορεία χρειάζεται κάποιος χρόνος και χρειάζεται και θάρρος, αν θέλετε, οραματισμού και πρόβλεψη κάποιων προκλήσεων. Η Παγκοσμία Τράπεζα ε, ανοίγει το δρόμο. Θα υπάρξει το σχετικό φόρουμ στην Ουάσιγκτον. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ανοιχτή στις νέες ιδέες και μπορούμε να συνεισφέρουμε. Και αν υπάρχει μεγαλύτερη ενθάρρυνση, αν δώσουμε και εμείς μεγαλύτερη ενθάρρυνση στην Παγκόσμια Τράπεζα, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να έρχομαι στη συζήτηση αυτή με εξαιρετικά φιλόδοξες ιδέες και με ανοιχτά μάτια και καρδιά. Γιατί διαφορετικά υπάρχει μεγάλη κίνδυνος απογοήτευσης και ε, μείωση των προσδοκιών. Το θέμα είναι πού θα ξεκινήσουμε. Το θέμα είναι καταρχά να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στην ενέργεια. Γιατί η πρόσβαση στην ενέργεια σημαίνει ότι όχι μόνο υπάρχει αυτή η πρόσβαση, αλλά ταυτόχρονα ότι η ενέργεια αυτή θα είναι αηφόρο και αποτελεσματική. Εάν δούμε τι πρόσφατε τάσει στι διάφορε χώρε με τι οποίε συνεργαζόμαστε, υπάρχει τεράστια αστικοποίηση αυτή τη στιγμή. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή αλλάζει όλο το μοντέλο του ενεργειακού κύκλου. Δεν είναι μόνο το θέμα, ε, αν θέλετε, παροχής ενέργειας σε αγροτικές περιοχές, αλλά και σε μεγάλα οικιστικά σύνολα. Επομένως, η κοινωνική διάσταση είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της όλης στρατηγικής. Αλλά ταυτόχρονα, πολύ σημαντικό, είναι τα σχέδια ε, τα επενδυτικά. Με 200 εκατομμύρια ευρώ που διαθέτουμε δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Υπάρχει ανάγκη να κάνουμε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Γιατί πιστεύω ότι το σήμα κατευθέν της Ευρώπης θα πρέπει να είναι η ΑΠΕ. Και με αυτό και με τις δυνατότητες που προσφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα μπορούμε να κάνουμε κάτι σημαντικό, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την παροχή ενέργειας, αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε να σας πω κάτι στα ουγγρικά, στο τέλος, ότι